κυβερνήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση θα αντιμετωπίσουν αύξηση του πληθυσμού του αστικού που αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ποσότητα ε, αποβλήτων που θα παράγεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνονται τώρα οι παρεμβάσει ενό λεπτού και θα περάσουμε στη συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων. Ε, εκθέσεων. Πρώτη είναι η έκθεση του Ρικάρντο Λάστρα για την αναπτυξιακή συνεργασία με τη Λατινική Αμερική. Ο εισηγητή έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, στα πλαίσια των τωρινών διαπραγματεύσεων για ένα νέο όργανο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη 2014-2020. Η έκθεση την οποία τώρα σας εισηγούμε θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Λατινική Αμερική δεν είναι δυνατόν και ούτε πρέπει να περιθωριοποιηθεί. Το μήνυμα της Κομισιόν είναι ξεκάθαρο. Πάρα πολλέ χώρε τη Λατίνική Αμερική έχουν πετύχει του στόχου του όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και παρόλα αυτά θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να θεωρηθεί ότι πια για αυτού η αναπτυξιακή βοήθεια. όμω από την άλλη μεριά ε, είναι αλήθεια ότι τώρα έχουμε ένα φραγμό, έχουμε ένα... Έχουμε μια τροχοπέδη γιατί υπάρχει πάρα πολύ ανισότητα. Έχουμε το 41% των φτωχών όλου του πλανήτη σε αυτή την περιοχή και εκεί έχουμε, το, έχουμε 52 εκατομμύρια τα οποία ζουν λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα και εκεί πέρα κάποιες από τις χώρες έχουν, υπάρχουν έλλειμμα διατροφή πάνω 20% και αυτή είναι μια άλλη, η άλλη πραγματοδομόνη για τη Λατινική Αμερική και σε αυτό το κοινοβούλιο και σε αυτό το χώρο θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι είναι σημαντικό όλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Λατινική Αμερική και θα πρέπει να είναι ισχυρή. Η Λατινική Αμερική θα πρέπει να μπορεί να δίνει τη μάχη για την ανάπτυξή τη. Και οπότε θα πρέπει γι' αυτό το λόγο εμεί να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα, γιατί μα χρειάζονται. Ε, γι' αυτό και εμεί δεν συμφωνούμε με τις ε, ριζοσπαστικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εκθεσή της, γιατί εκεί πέρα θέλει να γίνει μόνο με οικονομικά κριτήρια ε, η διάκριση και θεωρεί ότι ο σημερινό, η Κολομβία και το Περού ε, δεν θα συμμετέχουν πια στην διμερή βοήθεια και επίσης συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνεργασία και την ενίσχυση της Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατία, η οποία ε, έχει πολύ καλύτερε επιδόσει, ε, αν όχι ίσε, με τι χώρε εκείνη τη Λατινική Αφρική. Οπότε αυτό είναι μια δεσμένη διάκριση βάρο τη Λατινική Αμερική. Ο, γι' αυτό και εμεί θέλουμε να γίνει μια διαφοροποίηση, θέλουμε να γίνει μια διάκριση με υπεύθυνο τρόπο, να έχουν υπόψη και άλλα κριτήρια, οι, οι και επίση να ληφθούν υπόψη και άλλοι συντελεστέ και άλλε μεταβλητέ. Οπότε και αυτού του είδου το μέσο πολιτική για την ανάπτυξη ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη χρήση τη φτώχεια και έτσι θα πρέπει να δώσουμε προστιθέμενη βοήθεια ε, από αυτήν την αναπτυξιακή βοήθεια και γι' αυτό θα πρέπει να θέσουμε σε ενέργεια μια ανάπτυξη για κάθε χώρα της περιοχής και έτσι να μεγιστοποιήσουμε την ε, ενίσχυσή μας, την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και έτσι να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο, πιο δυναμικό μας το μήνυμα προς τους φίλους εταίρους της Λατινικής Αμερικής. Αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει είναι να δούμε πώς θα παγιωθούν τα επιτεύγματα, τα οικονομικά και κοινωνικά της περιοχής εκείνης, να εστιάσουμε εκ νέου την προσοχή μας ε, και να έχουμε συνευθύνη για όλες αυτές τις χώρες και έτσι να μπορέσουμε να τους δώσουμε την, ε, να τους δώσουμε την, την, την ενθάρρυνση για να έχουν καινούργιες πολιτικέ, πολιτικές, ε, να προχωρήσουν προ νέα τεχνολογία, νέα ενέργεια, ε, να καταπολέμψουν την ανασφάλεια του πολίτη και μια σωστή πολιτική που να στέλνει του πόρου του πιο ευάλωτου και σε αυτή την έκθεση αυτό το οποίο ζητείτε είναι να συνεχιστεί η πολιτική της ενίσχυσης και οποιαδήποτε περικοπή των πόρων ε, να μην αφορά τους ε, πιο ευάλωτους της χώρας. Επομένως, προσοχή γιατί 11 χώρες κόβονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη διμερή συνεργασία. Άρα, δεν συμφωνούμε με αυτή την άποψη, τη θεωρούμε πάρα πολύ ζωσπαστική και θέλουμε να γίνει ένας επαναπροσανατολισμός αυτής, αυτού του, του, του, μέσου πολιτικής για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιγητά. Θα ήθελα ε, να ρωτήσω αν έχετε μια μπλε κάρτα ή το catch the eye. Θέλετε να μιλήσετε στο πλαίσιο της διαδικασίας catch the eye. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κόρτες ε, Λάστρα για αυτή την εξαίρετη έκθεσή του. Η Λατινική Αμερική είναι μία από τις περιοχές του κόσμου και έχουν γνωρίσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την εξέλιξη και δεν είναι δεδειγμένη στιγμή για να αποσυρθεί η βοήθεια αυτή ξαφνικά. Αυτό θα πρέπει να γίνει βαθμιαία, ούτω ώστε να μπορέσουν οι χώρες αυτές να πηγιώσουν το κράτος δικαίου και να μειώσουν τους αριθμού της φτώχειας. Είναι σημαντικό να υπάρξει συνέχιση τη παροχής βοήθεια στι χώρε τη Λατινική Αμερική γιατί ε, οι χώρες αυτές παρόλο που έχουν ποσοστό ανάπτυξη της τάξης του 4% έχουν τεράστια ποσοστά φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική συμμερίζονται κοινέ αξίε και θα πρέπει να προχωρήσουν από κοινού, ώστε να αντιμετωπίσουν τι παγκόσμιε προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίε μα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, που υπάρχει μια παγκόσμια διαπλοκή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιράν... Ε, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Κόρτες Λάστρα και θα ήθελα να πω ότι ε, δεν θα πρέπει να περιορίζουμε την προσοχή μας στις οικονομικές πτυχές ανάπτυξης της Λατινικής Αμερικής. Εμείς θα προτείνουμε μία πρόταση η οποία ε, αντιβαίνει στα, στην παροχή ε, ε, βοήθειας προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εάν την αντικρίσουμε με άλλα μάτια μια στιγμή όπου ακριβώς μας δίνει εξαιρετικά δείγματα ανάπτυξης κοινωνικής προόδου, νομίζω ότι θα πρέπει να τη βοηθήσουμε ούτως ώστε να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Θα πρέπει να θυμηθούμε όλα τα επιτεύγματα επίσης σχέση με τον αυτόχθονα πληθυσμό των Ιθαγενών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φερέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρα. Στη Λατινική Αμερική σήμερα γίνεται μια διαδικασία εκπληκτική ε, που προξενεί ενθουσιασμό. Υπάρχει μια οργάνωση καλύτερη και κατάφερε τελικά η περιοχή να πετύχει την προόδο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι λογική οικονομική ανάπτυξη παρά την παγκόσμια κρίση, μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυξάνονται τα κοινωνικά δικαιώματα. Πρέπει όμως να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κενά. Υπάρχουν νέες προκλήσεις, νέες ανάγκες όσον αφορά την συνεργασία για την ανάπτυξη. Σε διάφορες χώρες χρειάζεται επαναπροσανατολισμός της συνεργασίας. Από ανάμεξη και πατερναλισμό θα πρέπει να περάσουμε προς οικονομική υποστήριξη και πολιτική υποστήριξη, συνεργασία για να απτυχθεί τεχνολογία και επιστήμη, σεβόμενη την κυριαρχία των λαών αυτών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα, ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε σχέση ακριβώ με την έκθεση που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό σε κάθε συμφωνία να θεωρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ε, βασική προϋπόθεση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερος όταν το ζητούμενο είναι ε, όταν ε, διακυβεύονται συγγνώμη τα δικαιώματα των πολιτών σε μια χώρα όπως είναι η Βολιβία όπου ε, ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, συνελήφθηκε κρατείται φυλακισμένος παρόλο που δεν οδηγήθηκε σε μια δίκαιη δίκη. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν δράση ώστε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επόμενο ομιλητή, ο κ. Σφαροβλάβ Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ. Η Λατινική Αμερική είναι μια περιοχή όπου υπάρχει μια συνεχής βελτίωση. Υπάρχουν παρόλα αυτά 180 εκατομμύρια πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις έδρες συνθήκες της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. Σήμερα συζητήσαμε για τη νέα πρόταση της ε, Επιτροπής, η οποία θέλει να αλλάξει το σύστημα γενικευμένων προεκτιμήσεων, κάτι το οποίο ενδεχομένως θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε αυτές τις ε, χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί. Είμαι πεπισμένος ότι μια κατάλληλη πολιτική η οποία θα συνοδεύεται από μια παροχή υλικής βοήθειας θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια θετική συνέχιση των καλών εξελίξεων στην Λατινική Αμερική. Κύριε Πρόεδρε, οι εθνικές οικονομίες της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν πληγεί τόσο από την δημοσιονομική κρίση. Το υπολογίζεται και μια ανάπτυξη τάξη του 4,5%. Ωστόσο, παρά τι ε, προγνώσει αυτέ, υπάρχουν 180 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο φτώχεια 10 ε, από τι χώρε της Λατινικής Αμερικής ε, συγκαταλέγονται μεταξύ των 15 όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερε ανισότητες. Επίση, υπάρχουν τεράστια ποσοστά εγκληματικότητα και βία κατά των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερο χορηγό, αλλά ο δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτή και οικονομικό εταίρο τη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε στην παγίωση του κράτου δικαίου αλλά και στην καταπολέμηση του προβλήματος της φτώχεια. Ε, γι' αυτό χρειάζονται ενισχύσει επιχειρήσεις ούτω ώστε να βοηθηθούν για ανάπτυξη και αυτοβοήθεια. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά σε αυτές τις εξελίξεις στην Ήπειρο αυτή. Ε, ε για αυτό το σημείο της αναπτυξιακής συνεργασίας με την Λατινική Αμερική ε, υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Όχι, λέει ο Πρόεδρος, άρα κύριε Επίτροπε, κύριε Τεχούχ, έχετε εσείς το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση έρχεται την πιο καλή στιγμή, διότι προσπαθούμε να εντοπίσουμε το μελλοντικό πλαίσιο συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε και τα βασικά θέματα των σχέσεων μα με τι χώρε της Λατινικής Αμερικής. Θα είναι σημαντική συνεισφορά αυτή στι συζητήσει για, για τα προτινόμενα εξωτερικά χρηματοστατικά μέσα και θα μπορέσουμε να καθορίσουμε στρατηγικές προτεραιότητες στην περιοχή. Έτσι, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι βασικές συστάσεις εκθέσεως εφηγραμμίζονται πολύ με τις τωρινέ και μελλοντικές απόψεις μας όσον αφορά τη συνεργασία με την περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Όπως λέει και ο συγητής, η Λατινική Αμερική έχει ετερογενείς χώρες, υπάρχει ποικιλομορφία ε, με διαφορετικές ανάγκες. Οι τελευταίες δεκαετίες έδειξαν τεράστιους μου ανάπτυξη στην περιοχή πολλές από τις χώρες μέσω εισόδημα έχουν τα αναγκαία μέσα και στέρεη βάση για να οικοδομήσουν διάφορα σχέδια εθνικής ανάπτυξης. Επανειλημμένα με προσέγγισαν διάφορες αναπτυσσόμενες χώρες που εξέφρασαν επιθυμία να απομακρυνθούν από προγράμματα ελάφρυνση μειώσεω των προβλημάτων στόχιας προς ανάπτυξη. Και με την ανακοίνωσή μα αυτό περιγράφουμε και με τα προτινόμενα χρηματοστικά εξωτερικά μέσα. Θα πρέπει να συζητήσουμε τους διαθέσιμους πόρους που χρειάζονται περισσότεροι πόροι που δεν είναι πολλοί και που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι πιο προχωρημένες χώρες θα βγουν από το πρόγραμμα ενίσχυσης και συνεργασίας. Αλλά θα κάνουμε άλλου είδους, θα δημιουργήσουμε άλλου είδους σχέσεις με αυτές τις χώρες για την ανάπτυξη. Θα διευκολύνουμε τις επενδύσεις, μέσω μηχανισμών ανάμειξης και περιφερειακών προγραμμάτων και υποφελούμενοι από την εμπειρία τους από τριμερή συνεργασία και από συνεργασία νότου-νότου. Για καλύτερη συνεργασία με τις προχωρημένες χώρες θέλουμε καλύτερα μέσα συνεργασίας που προτείνονται να ανεβάσουμε επίπεδο συνεργασίας, με άλλα λόγια. Ανεξάρτητα από την διαφοροποίηση των διαφόρων μέσων συνεργασίας, προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει αρκετού πόρους στη Λατινική Αμερική. Στα πλαίσια του μέσου ανέφερα, που σε συνδυασμό με τα διάφορα άλλα μέσα και προγράμματα θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε την καλύτερη στρατηγική για κάθε χώρα της περιοχής. Και αυτό σύμφωνα με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να ακολουθεί συνεχτική πολιτική για την ανάπτυξη, όπως αναφέρεται και στην έκθεση. Όσον αφορά τον καθορισμό των στρατηγικών, εντοπίστηκαν προτεραιότητες στην έκθεση. Αυτές οι προτεραιότητες ταιριάζουν με τις δικές μας. Παράρτημα 4β της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Μέσα Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Κλείνοντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει ενεργά να κινείται στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Όμως οι σχέσεις μας με την περιοχή οριμάζουν. Άλλαξαν. Από σχέση δωρητού αποδέκτου ε, φτάσαμε σε ισότιμη βάση. Τα προτινόμενα εξωτερικά μέσα θα μας δώσουν επαρκή ευελιξία και πεδίο. Ταυτόχρονα, σωστή συγκέντρωση και εστιασμό για αποτελεσματικές θετικές συνεργασίες με κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τι ούτω τρόπο. Βασιζόμαστε σε συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προσπάθεια που καταβάλουμε και χαιρόμεθα διότι η έκθεση αναγνωρίζει παρόμοιες προκλήσεις και προτεραιότητες όπως και εμείς.